Άρχεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως έχουν ήδη διανεμηθεί, δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις από ό,τι βλέπω, επομένως θεωρούνται εγκεκριμένα.